Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Σας παρακαλώ καθίστε. La séance est reprise. Συνεχίζουμε. Les votes sur le projet... Ψηφίζουμε για το σχέδιο προπολογισμού 2017. Θα ξεκινήσουμε με την εξέταση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου τμήμα 1. Έπειτα τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και κατά τρίτον τις πληρωμές. Donc je vous invite à vous saisir. Παρακαλώ να κοιτάξετε τα, τους φακέλους σας και να πάρετε τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου στα χέρια σας. Le premier amendement a pour objet Η πρώτη τροπολογία έχει στόχο να παραμείνει στο ίδιο μέγεθο ο προπολογισμό που εγκρίθηκε την Άνοιξη, υπέρ αυτή τη τροπολογία. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η δεύτερη για ε, τροποποιητικές ε, τροπολογίες μόνο ε, για επιπλέον πληρωμές θα γίνονται δεκτές, δηλαδή εξίσωση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Τροπολογίες Τροπολογίες 791, 791 ε, και 7198. Τις ψηφίζουμε μαζί από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Οι τροπολογίες περνούν με 21 ψήφους υπέρ και 15 κατά. Κύριε Γκάγερ, θέλετε το λόγο. Nous avons maintenant à Ο μπλοκ τώρα. 7089 και 7092. Υπέρ. Κατά. Amendement 2000... 2002. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέρας. Εγκρίνεται 27 προς 9 για 4 αποχές. Ψηφοφορία και πάλι ο μπλοκ μάλλον. Τροπολογίες 7.000 4.623, 4.656, 7.837 και 7.091 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7.285 ε, υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 1004. Υπέρ. Με συγχωρείτε. 7.981. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.404 και 4.836 υπέρ κατά απορρίπτεται. 7.835 και 4.821 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7.230 297 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7.839 και 4.821 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Να ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται 29 προς 11. 7.840 και 4.826 υπέρ. Κατά αποχές απορρίβεται. 7.303. Ε, υπέρ, κατά, να επεληθεύσουμε για δεν όλοι το χέρι τους. 7.303. Ε, Πέρας. Απορρίπτεται 33 προς 5. Παρακαλώ να σκόνετε τα χέρια σας. Τα 1841 και 4.327 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8.202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7.842, 4.628 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.629 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.630 υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 27 προς 15. 7.308 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιφυλάξεις. 4.246 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8.203. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8.205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παρατήρηση. 8.196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8.187 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.902 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7.843 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7.844 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71-96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71-97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71-99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και τώρα τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις. Γενικέ εισηγητά, θέλετε να μας επιβεβαιώσετε ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το γεύμα καταφέρατε να βγάλετε άκρη. Έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, έχουμε προσεγγίσει την ε, τελειότητα, αλλά δεν την έχουμε επιτύχει πλήρω. Ε, αν πάμε στη σελίδα 4, πάνω πάνω, υπάρχει μία... Το μέτρο 1, 2, 5 76 της Περιφερειακής Επιτροπής και από το ΕΛΚ. Αυτή η δράση ε, δυστυχώς περιλαμβάνεται δύο φορές στο κατάλογο, οπότε οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές μπορούν να ανέβουν από 500.000 στο 1 εκατομμύριο. Είναι λάθος αυτό. Οπότε αν το διορθώσουμε πλησιάζουμε στην τελειότητα. Τέταρτη σελίδα λοιπόν έλεγα, προπαρασκευαστικά μέτρα, ρέγγι, ε, 65-76 για τις περιοχές που υστερούν υποχρεώσεις και πληρωμές μπορούν να τις ε, ε αυξήσουμε από 500.000 στο 1 εκατομμύριο. Οπότε λίγη αυτό το θέμα. Αυτό που μας λέτε δηλαδή είναι να δεχτούμε και τι δεσμεύσει και τι πληρωμέ. Από 900.000 σε ένα εκατομμύριο. Αυτό λέτε κύριε Σιγητά. Πολύ ωραία. Άρα, ο κατάλογος που έχουμε μπροστά μας, όπως τροποποιήθηκε για τη γραμμή που αντιστοιχεί στην τροπολογία 6.576. Αντί για 900.000 φτάνουμε 1 εκατομμύριο. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν το έγγραφο συνολικά, όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Υπέρ του καταλόγου, όπως τροποποιήθηκε. Κατά. θες Ο κατάλογος εγκρίνεται. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Ε, στη γραμμή 020170 ε, και ψηφίζουμε μια σειρά από τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έχουν αποσυρθεί οι υπόλοιπε τροπολογίε, οπότε ολοκληρώσαμε με τι προφορίε για τι πιλωτικέ δράσει, για τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσει. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο τμήμα, πληρωμέ. Μισό λεφτάκι. Ωραία αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν ε, ψηφίσουμε για τις πληρωμές, να σας ε, ενημερώσω ότι υπάρχει μια τροποποίηση για τις ψηφοφορίες που κάνουμε σήμερα το πρωί στην τροπολογία 52-98 της ΑΦΕΤ για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, το τμήμα 10 του σημείο 4 δεν παρουσιάζει καθόλου πληρωμέ. Επειδή είναι μη διαχωριζόμενε δαπάνε, θα πρέπει να εισαγάγουμε εκεί τις πληρωμές που αντιστοιχούν στις, δεσμεύσει, στις υποχρεώσει. Το ποσό είναι 800.000 ευρώ. Θα γίνει αυτή η τεχνική τροποποίηση. Για τις πληρωμές τώρα. Έχουμε δύο μπλοκ τροπολογιών. Το πρώτο αφορά την επαναφορά την επαναφορά του επίπεδου των πληρωμών που περιέχονται στην πρόταση της Κομισιόν ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα είναι υποτροπολογία που βλέπετε μπροστά σας να ξεκινήσουμε με αυτήν την υποτροπολογία ή να ψηφίσουμε συνολικά το μπλοκ, το δεύτερο αυτό μπλοκ, και είναι τμήμα του και η τροπολογία για τα 5 εκατομμύρια. Είναι συστατικό του τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη ε, έτσι τροποποιημένη τροπολογία. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται και αυτό το δεύτερο μπλοκ. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλήξαμε με τις ψηφοφορίες για το σχέδιο προϋπολογισμού 2017. Για άλλη μια φορά να συγχαρώ τον γενικό μας εισηγητή και όσους συνέβαλαν. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συνεργάτες μας και ελπίζω ότι ο διάδοχος της κυρίας Γεωργίεβα θα στηρίξει τις προτάσεις μας, θα σεβαστεί τις ψήφους μας. Και ελπίζω το Συμβούλιο να επιδείξει και πολύ κατανόηση. Ευχαριστώ τον κύριο Ταγάν για τα άλλα τμήματα και εκείνος για τα υπόλοιπα τμήματα επέδειξε αποφασιστικότητα, συνέπεια. Ας πιστέψουμε στο όνειρο ότι όλες μας οι τροπολογίες θα γίνουν δεχτές από το Συμβούλιο όταν θα έρθει η ώρα της συνδιαλλαγής. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τελειώσαμε. Έχουμε ακόμη πολλές εκθέσεις. Όσοι θα ήθελαν να αποχωρήσουν, παρακαλώ να αποχωρήσουν ησύχως και συντόμως για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ησύχως παρακαλώ. Okay. Ναι. βρήκαμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να κάνω απολογισμό αυτού που μου αναθέσατε για τη γενική αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού του σώματος. Κοιτάξτε. Σταματήστε παρακαλώ να θορυβείτε στους διαδρόμους, ιδιαίτερα από τη δεύτερη σειρά και μετά, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα. Όσοι θέλουν να φύγουν, παρακαλούνται να το φύγουν, να το πράξουν. Ταχαίως. Λοιπόν, μου είχατε ζητήσει να γίνουν κάποιες τροποποίησεις του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Το πλαίσιο είναι η πείρα που συλλέξαμε και κυρίως οι εισηγητές μας. Οι εισηγητές μας που ήταν εισηγητές για τον προϋπολογισμό Ντεπρέ 16 και Τάραν για το 17 και ιδιαίτερα για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου ο οποίος ξέρετε, οδήγησε σε παρανοήσει και έλλειψη κατανόηση. Η ΑΦΚΟ, με εισηγητή τον συνάδελφο κ. Κόμπετ, κάνει επίση προτάσει για τροποποίηση του ιστορικού κανονισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απόλυτα λογικό να συμβάλλει και η δική μας Επιτροπή. Σημειώνω ότι μια ομάδα εργασία με κεφαλή στον αντιπρόεδρο Βίλαντ οργάνωσε διαβουλεύσει διοικητικού τύπου για να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του εσωτερικού μας κανονισμού. Η πρόταση που θα σας κάνω χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ένα τεχνικό τμήμα και ένα τμήμα που θα το χαρακτήριζα πιο πολιτικό. Για το τεχνικό πρώτα απ' όλα τμήμα. Σας προτείνω να κάνουμε τις ε, διαδικασίες εξοχολογισμού του κανονισμού που είχε υποβάλει και η ε, η ομάδα εργασία Βίλαντ, ε, τροπολογία 3 για τροποποίηση του άρθρου 95 για να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητε και ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων badge και κοντ. Επίση θα σας πρότεινα να επιμείνουμε επί τις αρμοδιότητές μας για τα ειδικά οχήματα, τα ειδικά μέσα. Ορισμένες φορές υπάρχουν ε, συγχύσεις και έλλειψη κατανόηση για αυτά τα ειδικά οχήματα και ειδικά μέσα. Άλλες επιτροπές ήθελαν να είναι αρμόδιες για τη λειτουργία. Τροπολογία 9 στο, παράδειγμα, 6 που αφορά ακριβώς τον εσωτερικό κανονισμό. Θα θυμάστε ότι η Λίμπη έχει επιχειρήσει να θεωρηθεί συναρμόδια για την κινητοποίηση ενός ειδικού μέσου για τους πρόσφυγες. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε σαφέστατα ότι όταν ε, διακυβεύονται ειδικά μέσα είναι αρμοδιότητα τη επιτροπή Προπολογισμών. Τώρα να περάσω στο τμήμα τροπολογιών που θεωρώ πιο πολιτικό και θεωρώ ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον για την Επιτροπή μα. Ασχολείται με την τροποποίηση του εσωτερικού λοιπόν με τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου, τη σχέση μα με το Προεδρείο και στα πλαίσια τη διαδικασία έγκριση του προπολογισμού υπήρξαν πολλέ φορέ διαφωνίε και απογοητεύσει το Προεδρείο εκπονεί ένα σχέδιο. Παίρνουν τη γνώμη μας, ε, συζητάμε μέλη του Προεδρείου, εισηγητέ και σκιώδεις, προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τις θέσεις μας, αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη της ε, έκβασης, γιατί θα είναι έκθεση μπάτζου που θα περάσει στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Και το Προεδρείο, σε τελευταία ανάλυση, κάνει αυτό που θέλει. Θυμόμαστε τι έγινε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια που αμφισβητούσε την επάνωδο εντός του υπαλληλικού σώματος των οδηγών και μετά, κάποια λεπτά μετά, ε, διαπιστώσαμε ότι έγινε μια προκήρυξη για πρόσληψη οδηγών ως εξωτερικών συνεργατών. Προτείνω τρία σημεία. Το πρώτο προσπαθεί να διευκρινίσει τις ευθύνες των μεν και των δε, τις αρμοδιότητες, να τις ε, διαχωρίσει και θέλουμε να είναι η τελευταία λέξη να ανήκει στη δική μας επιτροπή πριν την Ολομέλεια, αν υπάρχει έλλειψη κατανόησης. Εάν αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη μιας δημοσιονομικής απόφασης, τότε πρέπει να έχουμε την πλήρη αρμοδιότητα για να αναλάβουμε αυτή την πολιτική ευθύνη. Προτείνω λοιπόν η κατάσταση προβλέψεων να εκπονείται από το Προεδρείο, να είναι αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής μας και ε, αυτή η έκθεση μετά τις αναγκαίες συνεννοήσεις και συμβασμούς να είναι η έκθεση τη οποίας θα ψηφίσει η Ολομέλεια. Θα υπάρξει φάση συνδιαλλαγής, ε, επιδίωξη συμφωνία, αλλά σε τελευταία ανάλυση θα είναι έκθεση Bunch. Τελικά λοιπόν, εμείς πρέπει να διαπραγματευτούμε το Γενικό Προϋπολογισμό με το Συμβούλιο, τη Δημοσιονομική Πειθαρχία από την οποία εξαρτάται και η αξιοπιστία μας έναντι των άλλων οργάνων. Διότι αν υπάρχουν υποψίες ε, χαλαρότητας, υποψίες έλλειψης σοβαρότητας στις σχέσεις μας με το Συμβούλιο, η αξιοπιστία μας ε, θα αμφισβητηθεί σοβαρά. Η δεύτερη πρόταση που διατυπώνω βασίζεται στην αρχή ότι Πρέπει να υπάρχει απέτηση μέσω προθέσμων και μακροπροθέσμων χρηματοδοτήσεων που να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των ε, δαπανών ε, επενδύσεων και των τρεχουσών δαπανών. Το είπαμε και στην έκθεση Τάραντ. Κάθε προπολογισμό θα πρέπει να γράφεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να μην πηγαίνουμε στα τυφλά. Χθε είδα μια έκθεση του Γενικού Γραμματέα όπου λέγεται ότι εφόσον εγκρίθηκε το Brexit δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Μια τέτοια απάντηση είναι απαράδεκτη. Και διαμαρτύρομαι έντονα έναντι αυτής της στάσης του Γενικού Γραμματέα. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Προτείνω ότι οι συνάδελφοί μας στο Προεδρείο όταν συζητιέται ο προπολογισμό να ζητούν να γίνεται ονομαστική ψηφοφορία για την κατάσταση προβλέψεων. Διότι πρέπει να εκφραστούμε και στην Ολομέλεια. Όταν υπάρχουν ονομαστικές πλειο, τότε προσέχουμε καλύτερα τι ψηφίζουμε. Ε, είναι βασικές παλιές αρχές ε, των υγιών και χρηστών δημοσιονομικών. Το άρθρο 15 της διακήρυξης ε, των δικαιωμάτων του πολίτη και του ανθρώπου λέει ότι η κοινωνία έχει δικαίωμα να απαιτεί λογοδοσία από οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό. Τα πρακτικά του Προεδρείου σήμερα εγκρίνονται με ευρεία, ε, συγγνώμη, Όπω λένε τα πρακτικά του Προεδρείου, τα περισσότερα στοιχεία της κατάστασης προβλέψεων ψηφίζονται με ευρεία πλειοψηφία. Νομίζω ότι οι ονομαστικές ε, ψηφοφορίες επιτρέπουν να καταλάβουμε καλύτερα πώ ψήφισε ο καθένα. Γιατί ορισμένε φορέ λαμβάνονται κάποιε αποφάσει και ρωτάμε κάποιου, μα τι ψηφίσατε και δεν είναι σε θέση να μα απαντήσουν. Έτσι νομίζω θα προσέχουν όλοι πολύ περισσότερο όταν συζητιέται ο προπολογισμό. Σας προτείνω λοιπόν αυτές τις ε, τροπολογίες είναι εννέα. Θα μας επέτρεπαν να καθορίσουμε τις αρμοδιότητες των μεν και των δε και να περικόψουμε και κατά ένα κανόνα τον ε, εσωτερικό κανονισμό. Όλες αυτές οι τροποποίησεις μπορούν να μπουν σε ένα άρθρο. Je souhaiterais entendre vos, vos observations, vos réactions. Monsieur Fernandez. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εργασία σας. Τώρα θέλετε να αντιδράσω έτσι αθερμό. Γιατί για τα θέματα αυτά εργάζονται διάφοροι. Θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη και αυτών των ατόμων. Τώρα είναι τόσο επίγον και θα ήθελα να μάθω αν μπορούν να τροπολογηθούν οι τροπολογίες σας. Είναι πρόταση για την επόμενη Ολομέλεια. Αρτσουή. Όχι, όχι. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων και βάσει αυτής και να δούμε και πώς θα πάνε και οι ψηφοφορίες για τον προβλησμό του 17. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να υπάρχει χρόνος και για τους ίδιους τους βουλευτές που τους είχε εκλέξει ο λαός, να μπορούν να μας πούν ανοιχτά τη γνώμη τους, να μας ανοίξουν την καρδιά τους. Τώρα θα κάνουμε μια ανταλλαγή υπόψεων. Στις 4 Οκτωβρίου στις 3 η ώρα θα λήξει η προθεσμία υποβολής τροπολογιών στην έκθεσή μου. Στις 11 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και στις 8 Νοεμβρίου θα ψηφίσει η ΑΦΚΟ. Κύριε Φερνάντες. Να σας ευχαριστήσω. Και εγώ. Να ε, δούμε λοιπόν τι τροπολογίε και κατά πόσο θα μπορέσουν να τροπολογηθούν και εγώ όπω και πρόεδρο, πάντα λέω αυτό που έχω κατά νου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικό το θέμα των πολιτικών συμβούλων, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουν άποψη τελικά οι βουλευτές. Ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο πρέπει να το ομολογήσουμε ότι έχουμε εξαιρετικού βουλευτέ. Και πολλές φορές οι πολίτε δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν είναι απολύτω ανήμεροι. Μην υπονομεύουμε δηλαδή και τη θέση μας και το ρόλο που διδραματίζουμε. Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε, για τη δουλειά σας. Είναι σημαντικά τα θέματα διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό να είναι και, παρηχαρακά, να είναι και σαφής η ρόλη όλων. Να υπάρχει λοιπόν διαφάνεια, να υπάρχει υπευθυνότητα, αλλά να... για να υπάρχει και υπευθυνότητα θα πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καρδία Σαμπάλα. Ναι, συγγνώμη πρόεδρε, ήμουνα σε άλλη συνεδρίαση ε, και καθυστέρησα λίγο και δεν είχα την τιμή να ακούσω την παρουσίαση της έκθεσής σας. Δεν ξέρω αν έχουν οι συνάδελφοι να κάνουν κάποια σχόλια και προφανώς θα τα εξετάσουμε και θα καταθέσουμε αν χρειαστεί τροπολογίες. Ο κ. Κόντολα. Ε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομο σήμερα. Μία μικρή τοποθέτηση, επιτρέψτε μου. Επί της αρχής, πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπατε. Τα υποστηρίζω. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω διπλά και τριπλά την ε, διαφάνεια που χρειάζεται. Ε, κατά ονομαστικές ε, μεταξύ άλλων για να μπορέσουμε να δείξουμε και στους πολίτες τι υποστηρίζουμε ως βουλευτές. Αυτό πραγματικά ε, επικρίνεται σήμερα και δικαίω ότι οι απόψεις ε, που προβάλλονται στην χώρα του καθενός ε, και στο εκλογικό κοινό του καθενός δεν είναι απαραίτητα αυτέ που στηρίζουμε εδώ στο Κοινοβουλίο. Χρειάζεται διαφάνεια λοιπόν. Συμφωνώ. Κάτι άλλο τώρα, το οποίο και εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό και συνάντηκα όπω με αυτά που είπατε. Πιστεύω ότι τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου είναι γενικά πολύ ογκώδη. Τίνουν να είναι πολύ ογκώδη. Και δεν μιλάω μόνο για την έκταση του κειμένου, αλλά και για το περιεχόμενο που καλύπτουν. Κάποιες εκθέσεις φτάνουν τα 50 έως και 100 σημεία, τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι πάντα απαραίτητα να αναφέρονται. Νομίζω ότι τα συνέτεινε προς τη διαφάνεια το να είμαστε πιο επικεντρωμένοι στα κείμενά μας. Να εκφράζει δηλαδή και ο ίδιος ο τίτλος του κειμένου το τι πραγματικά πραγματεύεται το κείμενο και έτσι νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών μας. Ναι, πάρα πολλές ε, πληροφορίες δηλαδή, αυτό εννοείται. Και αυτό προφανώς ε, δεν συμβάλλει στην διαφάνεια του κειμένου. Ο κύριος Ντεπρέα. Euh, Δεν είμαι πλέον ε, εισηγητής, πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Ναι, αλλά για την εκτέλεση. Να πω ότι εκτιμώ τη δουλειά σας όχι μόνο γιατί έχει περισσότερη διαφάνεια, αλλά και σαφήνεια στο πώς ε, διαμορφώνεται η αλληλουχία των ε, διαφόρων ενεργειών και πώς θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών για το σχέδιο προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Προσωπικά βρίσκω ότι οι τροπολογίες, κατά τη δική μου την άποψη, η ε, πιο σημαντική από όλες αυτές είναι η πέμπτη. Στην τροπολογία 5 δίνετε τον ορισμό ε, για την διαδικασία που καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθενός. Οπότε πιστεύω ο εισηγητής, ε, το Προεδρείο μάλλον, μπορεί να εγκρίνει την πρόταση, διότι το Προεδρείο δεν είναι απλώς ε, ένα βοηθητικό όργανο του Γενικού Γραμματέα, αλλά μπορεί να εγκρίνει δικέ του προτάσεις. Όλα αυτά σωστά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού και μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Το βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικό διότι έτσι έχουμε μία έποψη για το τι θα συμβεί και μελλοντικά τα επόμενα χρόνια. Και επίσης, ξέρω ότι αυτή η ιδέα σας είναι ιδιαίτερα προσφυλής, η πρόταση όπως διατυπώνεται κάνει μια σαφή διάκριξη μεταξύ του εκτελεστικού προπολογισμού, δηλαδή τα έξοδα λειτουργίας και τις δαπάνες για επενδύσεις. Συμφωνώ με τις ε, περισσότερε λοιπόν τροπολογίε που Η έκτη τροπολογία διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα και την ε, αναπομπή στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ένα μικρό ερώτημα, μια απορία για την υποχρέωση που αναλαμβάνεται να έχουμε ονομαστική ψηφοφορία εντός του Προεδρείου. Καταρχήν, παρά είναι διαφανές ε, το σύστημα. Δεν έχω κάτι εναντίον της διαφάνειας. Όμως, με τον κανονισμό που εγκρίναμε θα περάσει αυτό ή με τον ιστορικό κανονισμό του Προεδρείου. Εσείς θα πρέπει να, να αποφασίσετε. Ε, θα αφήσουμε στο Προεδρείο την ελευθερία να ε, εγκρίνει τους κανόνες βάσει των οποίων θα αποφασίσει για διάφορα πράγματα. Αυτό ε, θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχω εγώ συγκεκριμένη άποψη, δεν έχω καταλήξει σε, κάποιο, σε κάποια τοποθέτηση, αλλά θα ήμουν κάπως πιο επιφυλακτικός από ότι ίσως εσείς και κάποιοι από τους συναδέλφους. Όχι γιατί θα ήθελα να είναι αδιαφανείς οι διαδικασίες, δεν είναι ότι θέλω η αδιαφάνεια να παραμείνει ο κανόνας, αλλά Πρέπει να σκεφτούμε πού ε, στο σύνολο των κανόνων μα θα βρούμε αυτή τη δυνατότητα για το Προεδρείο να μπορεί να οργανωθεί και να λαμβάνει ελεύθερα τι αποφάσει του. Εγώ δεν έχω προκαθορισμένη απάντηση, δεν έχω καταλήξει. Απλώ θέτω το ερώτημα. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Φερνάντε. Σα ακούω και σα παρακολουθώ. Δεν έχω το έγγραφο μπροστά μου Καταλαβαίνω όμως ότι άλλοι το έχουν ήδη στα χέρια τους, εμείς πάντως δεν το έχουμε. Οπότε δεν μπορώ να ε, πάρω θέση. Και μάλιστα επί της ουσίας για μια δήλωση προφορική χωρίς έγγραφο μπροστά μου. Είναι σημαντικός βέβαια ο διάλογος. Και θα μπορούσαμε να το ξανασυρτήσουμε σε σχέση με τα recall vote Για τις ονομαστικές λοιπόν ψηφοφορίες, γιατί κάποιοι πιέζουν, πιέζουν και λένε ότι στον τύπο ακούγονται πολλά για τα δίκτυα, του πώς ψηφίζουμε, τα κυκλώματα μάλλον, για το πώς ψηφίζουμε και ότι πρέπει επίσης οι βουλευτές να έχουν ελευθερία για να αποφασίζουν ε, όπως θέλουν και αυτό είναι κάτι βασικό. Πρέπει να τα σκεφτούμε. Αλλά αφού δούμε το έγγραφο Ευχαριστούμε κύριο Στάρεν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και νομίζω ότι αυτά που συζητάμε τώρα εδώ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουμε μπροστά το γραπτό κείμενο, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε λοιπόν εδώ και δύο χρόνια στην Επιτροπή Προπολογισμού και Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Η αρχή του προϋπολογισμού είναι στην αρμοδιότητά μας, θεωρητικά, αλλά ουσιαστικά άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις αντί για εμάς. Και εμείς, τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού, τελικά φέρουμε ευθύνη για αποφάσεις που έχουν λάβει άλλες ομάδες, άλλα άλλοι άνθρωποι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή. Αλλά να σας πω ότι στην τελευταία θετία, το 2009 στο 2014, ήμουν μέλος της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων. Και πραγματικά ήταν πολύ οδυνηρή η εμπειρία αυτή. Γιατί με πολύ αργό τρόπο α, καταλήξαμε στις νέους κανον... πρώτες γραφές του κανονισμού για τέτοιες προτάσεις λοιπόν τις οποίες καταθέσαμε ε, στην Ολομέλεια. Τελικά αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Ήταν σημαντικά λοιπόν τα ζητήματα αυτά. Τώρα λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι υπάρχουν τρία στοιχεία. Το ένα το έδειξε εδώ και καιρό το έχει θίξει ο πρόεδρος Αρτουή ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των λειτουργικών εξόδων και των στρατηγικών επενδύσεων. Υπάρχει ε, το σημαντικό θέμα του χρονοδιαγράμματος, ποιος προτείνει τι και σε ποια χρονική φάση και πότε πρέπει να απαντήσουν ε, τα, το κάθε θεσμικό όργανο. Και Ύστερα υπάρχει και το θέμα της ευθύνη. Θα ήθελα να υποστηρίξω την ιδέα του Πρόεδρου για την ονομαστική ψηφοφορία. Θεωρώ ότι ενδεχομένως να αποτελεί καλύτερο τρόπο. Να ξέρουμε ε, ποιος είναι υπεύθυνο για ποια ψήφο. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε στο Προεδρείο τι κανόνες θα ακολουθήσει και πώς τη συμπεριφορά θα ακολουθήσει στις συναντήσεις του. Αλλά από την άλλη, οι συνάδελφοι σύντομα, όπου να είναι, ξέρετε, θα εκλέξουμε το νέο πρόεδρο. Νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να αποστείλουμε ένα μήνυμα. Αυτά είχα ουσιαστικά να σας πω. Για το θέμα. Αλλά θεωρώ ότι ως Επιτροπή θα πρέπει να κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες, αλλά σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, θα μπορέσουμε να περάσουμε τα σημεία αυτά μόνο αν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του προπολογισμού του 2014 παρά τον ε, Φάραντς και την ε, Λεπέν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργούσε ακόμα και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα σωστό βήμα για τη βελτίωση του κανονισμού. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Ευχαριστώ, κύριος Γκυγιό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγκάια. Ναι. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το κείμενο πλήρω. Έχετε κατανόηση, βέβαια. Τι τελευταίε μέρε ήμουν απόλυτα αφοσιωμένο στον προπολογισμό. Άκουσα αυτά που είπατε, αλλά θέλω να κάνω μια θεμελιώδη παρατήρηση. Αρμοδιότητα της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι να προετοιμάζουμε ως ειδική την εργασία της Ολομέλειας. Όταν πρόκειται για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, δεν είμαστε μόνο κάποιοι που είναι πάνω από το Προεδρείο. Διότι το Προεδρείο είναι το Προεδρείο. Σε τελευταία ανάλυση αυτοί φέρουν την ευθύνη για την εκτέλεση του προπολογισμού. Και ως ειδική επιτροπή έχουμε συμβουλευτικό ρόλο βεβαίως. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτός μας ο ρόλος μας επιτρέπει να αγνοήσουμε, να διορθώσουμε ή να καταργήσουμε αποφάσεις του Προεδρείου. Έτσι είναι η, η λογική της δομής του Κοινοβουλίου. Τώρα για το θέμα ονομαστική ή όχι, άκουσα τι είπατε, αλλά σε τελευταία ανάλυση η ονομαστική ψηφοφορία αν είναι τόσο σαφής ε, που να είναι 15 υπέρ 0 ε, κατά είναι σαφές το αποτέλεσμα Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της επιστροφής εντός ε, της υπηρεσίας των οδηγών της κατάργησης δηλαδή της ιδιωτικοποίησης τι σχέση έχει αυτό Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού εργάζεται πολύ σκληρά να λαμβάνουμε πληροφόρηση όταν κάνουμε απαλλαγή για το Συμβούλιο να λαμβάνουμε πληροφόρηση για το πώς εκτέλεσαν τον προπολογισμό τους. Και δεν τη λαμβάνουμε γιατί υπάρχει λέει μια συμφωνία κυρίων από τη δεκαετία του 70 που λέει τότε που βέβαια ήταν διαφορετικός ο θεσμικός συσχετισμός δυνάμεων. Υπάρχει μια συμφωνία λοιπόν έλεγα που λέει ότι εμείς δεν κοιτάμε τόσο πολύ στο εσωτερικό του προπολογισμού του Κοινοβουλίου και αντίστροφα το Κοινοβούλιο δεν κοιτάει τόσο πολύ στο εσωτερικό του δικό μας προπολογισμού. Αν χρησιμοποιήσουμε όμως αυτή τη λογική τότε θα έχουμε προβλήματα αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την λογική έναντι τους κομισιών. Αν το κάνουμε κάτι τέτοιο, επειδή είναι το άλλο σκέλος της αρχής επί του προπολογισμού, θα θεωρήσει ότι θα έχει πολλές δυνατότητες να εξετάσει από κοντά το δικό μας ε, προϋπολογισμό. Να μην εκτεθούμε λοιπόν σε αυτό το κίνδυνο Να μην κάνουμε προτάσεις που μπορεί να είναι παράτολμες και τις οποίες ε, μπορεί μετά να αξιοποιήσει το Συμβούλιο για να μπει στα εσωτερικά μας και να κοιτάξουμε πολύ κοντά τα εσωτερικά μας. Δεν νομίζω είναι κάτι που θα το θέλαμε αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Ο κύριος Ντεπρέ. Πρόεδρε, δεν θέλω ακριβώ να κάνω παρέμβαση. Μια ερώτηση θέλω να απευθύνω στον κύριο Γκάγερ. Πραγματικά καθόλου δεν βλέπω πώς οι προτάσεις που διατυπώνονται εδώ θα επιτρέψουν στο Συμβούλιο, το οποίο δεν ανηφέρεται στις προτάσεις εδώ, θα επιτρέψουν στο Συμβούλιο να παρηθέσει. Δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στο ότι θέλουμε να ε, επηρεάσουμε τι δαπάνε του Συμβουλίου, όπω το ίδιο κάνει και το Συμβούλιο. Δεν ασχολείται με τι δαπάνε του Κοινοβουλίου. Τώρα για τη μείωση 5% αυτή γίνεται γιατί αναφέρεται στην διαθεσμική συμφωνία, όπω ε, την ε, ε, προσυπέγραψαν και τα τρία θεσμικά όργανα και μεταξύ μας συμφωνούμε για να προχωρήσουμε στις ανάλογες μειώσεις. Τώρα δεν μπορεί να έρθει το Συμβούλιο να πει στον επίπεδο των συνεργαστών μας ότι θέλω ε, να διαφωνήσω και θα βγάλετε τόσες θέσεις από το ΕΛ και από τους σοσιαλιστές. Δεν έχω δει πώς θα ψηφίσουν οι φιλελεύθεροι. Νομίζω ότι είναι θετικό το πρόσημο. Οπότε, ε, Ζωζέ, η κακή πίστη δεν είναι ποτέ επιχείρημα. Ναι, αλλά εγώ μιλάω εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Δεν ε, θεωρώ ότι είναι κάποιο άλλο αρμόδιο για να το κάνει. Εάν με επιτρέψει έτσι, δεν θα μιλήσει εσύ για την ομάδα μου. Παρά το σεβασμό που σου έχω. Ναι, παρακαλώ να μην μιλάτε ταυτόχρονα για το λόγο και ο κύριο Ντεπρέ. Λοιπόν, ε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκάγερ προ το εξή. Το πρόβλημα των ονομαστικών ψηφοφοριών, των ηλεκτρονικών. Νομίζω ότι αυτός αυτό το σύστημα κανόνων έχει ένα χαρακτήρα κάπως καχύποπτο και μάλιστα τιμωρητικό, διότι πολλά παραπέμπονται στα πρακτικά. Νομίζω, Πρόεδρε, το πάτε, την πάτε λίγο μακριά τη βαλίτσα εδώ πέρα, αλλά πραγματικά εδώ θα ε, αναφέρω πάλι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί να περιληφθεί αυτό το σύνολο των κανόνων. Το Προεδρείο βλέπω να δυσκολεύεται να το αποδεχτεί και νομίζω ότι όλο αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από τη λύση. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Φερνάντε. 30 δευτερόλεπτα. Απλώς να πω ότι συμφωνώ με την παρέμβαση του Ζεράρ. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μιλήσω εξ ονόματος του ΕΛΚ Εάν ε, προσέθετα για τους φιλελεύθερους, πραγματικά θα έπρεπε να σοπάσω τελείως. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Και για τους δύο. Δεν μιλάω για την ψηφοφορία, μιλάω για τη γένεση της πρότασης. Κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάω για τη γένεση της πρότασης και καθόλου για την ψηφοφορία. Έλεγα πώς ε, έφτασε αυτή η πρόταση των 76 θέσεων να πάρει σάρκα ε, ναι, είναι πραγματικά αξιοπερίεργη. Και καλό είναι να πάρουμε και πολιτική θέση, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι γενικοί γραμματεί των ομάδων ε, καθορίζουν το τι θα κάνουμε εδώ σε αυτό το σώμα και αυτό δεν μπορώ να το παραδεχτώ να το αποδεχτώ. Αν έχω κάτι να καταλογίσω στην ομάδα μου είναι ότι δεν υπήρξαν συζητήσει γι' αυτό. Λέμε, ε, καλά οι υπόλοιποι θα συμφωνήσουν αφού προτείνουμε αυτό. Τι είναι όλα αυτά, έτσι θα ζώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι θα ζώσουμε την εικόνα μια δημοκρατία που είναι διαφανή. Σε καμία περίπτωση. Εδώ πραγματικά ε, απειλούμε του ίδιου του εαυτού μα με τέτοιε στάσει και πραγματικά θα θέλει οι πολιτικέ ομάδε να αναλάβουν ξανά τι ευθύνε του. Προηγουμένω δεν ψήφισα για τι 76 θέσει εργασία διότι είχα κορεστεί από τις ε, αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, αλλά στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου πραγματικά θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Είχα τοποθετηθεί και την περασμένη φορά και θα πρέπει να πάρουμε θέση. Δεν τα ξαναπώ. Λοιπόν, ε, για τις ονομαστικές ψηφοφορίες, ναι, το πήγα λίγο μακριά, αλλά εάν ξεκινήσουμε να αυτολογοκρίνουμε τις προτάσεις μας, ε, θα καταλήγουμε σε συνενέσεις ε, χωρίς καμία προστιθέμενη αξία. Θα έλεγα τουλάχιστον ε, μετρία ε, ποιότητα. Πραγματικά λοιπόν, ναι, θέλω να την πάω πιο μακριά τη βαλίτσα. Γιατί κάποιε φορέ ευνηδιάστηκα όταν έμαθα το Προεδρείο το ψήφισε αυτό και το έδειξε στην αντιπρόεδρο τη ομάδα μου και δεν ήμουν βέβαιος. Μου είπαν ότι αυτό μπορεί να το δεχτούμε έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν είναι έτσι. ή Το κύριο μας έχει να κάνει με το πώς εμείς εδώ διαχειριζόμαστε τα δικά μας τα κονδύλια σε αυτό το ίδιο το κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το κύριο μας ε, εξαρτάται από το κατά πόσο δίνουμε το παράδειγμα, όχι μόνο από τα όσα λέμε και με το πόσε σελίδε έκταση έχουν οι εκθέσει. Θα μπορούσαμε να έχουμε κείμενα δύο σελίδων και να είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα γίνονται και κατανοητά. Το έκαναν ο κ. Μπακιά και η κυρία Μπερέ για τον προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Σε δύο σελίδε για να είναι εύληπτο και κατανοητό στου Ευρωπαίου πολίτε. Για να μην μιλάμε μόνο με εμπειρογνώμονες των νομικών. Με συγχωρείτε, αλλά έχω κι εγώ πραγματικά μια αφοσίωση στην αποστολή μου και στη θητεία μου. Κύριε Μπέγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχετε διαβάσει ακόμα το τελικό κείμενο, γι' αυτό μιλάτε. Το τελικό κείμενο το οποίο θεωρώ είναι αρκετά ρεαλιστικό σε κάθε φορά κάποια στοιχεία και θα πρέπει να το διαβάσουμε. Κοιτάξτε, τώρα για τις σκέψεις αυτές που μου αναφέρατε. Ακούσαμε πολλά σωστά επιχειρήματα για την διαφάνεια, για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί και ο τρόπος που ακολουθούνται οι διαδικασίε εδώ στο Κοινοβούλιο, τα είπε και ο κ. Σταράντ. Και τα έχουμε σχολιάσει επισταμένως αυτό και ε, στην Επιτροπή, ότι κάποια έγγραφα της διοίκηση σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι είναι πολύ καθυστερημένη η άφηξη των εγγράφων αυτών εδώ στην Επιτροπή και δεν είχε χρόνο ουσιαστικά ο εισηγητής να τα εξετάσει λεπτομερώς. Πέρα από το θέμα της ονομαστικής κλίσης, εγώ δεν έχω ιδιαίτερα πρόβλημα να αναφέρομαι κάπου στα πρακτικά. Τώρα κατά πόσον ε, αυτό θα βοηθήσει τις ε, ψηφοφορίες δεν ξέρω. Αλλά σε ό,τι αφορά την υπευθυνότητα και την ευθύνη που φέρουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, και σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των ομάδων, θα πρέπει να δούμε ποιον ε, εκλέγουμε στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Και αν εκλέγεται ο καθένας ε, επειδή ε, καταφέρνει να αντιεκπαιρεώνει υποθέσεις γρήγορα γρήγορα, όπως τα λέει η διοίκηση. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ. Ή κατά πόσον στο Προεδρείο και εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών πραγματικά εκτός πια αν υπάρχει κάποια κατεπίγουσα ανάγκη. Απορρίπτουμε τις ε, μεταφορές και τις προτάσεις αυτές αν δεν έχει διατεθεί το εκάστοτε κείμενο μία εβδομάδα ε, εκ των προτέρων στις ομάδες προκειμένου να έχουμε χρόνο να κάτσουμε να τα μελετήσουμε όλα αυτά. Όχι τελικά να χανόμαστε σε αριθμούς και παραρυθμούς και τελικά να χάνουμε την ουσία του θέματος. Και αυτά λοιπόν τα θέματα θα πρέπει να κάτσουμε να τα σκεφτούμε, πιστεύω, Πρόεδρε. Μπορεί κάτι να όριζε ο κανονισμός. Η Γκρέσλε είπε ότι και στα θέματα, στον κανονισμό του προπολογισμού αναφέρονται διάφορα στοιχεία, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις με νομική και δημοκρατική ευθύνη. Προ την κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα πρέπει να κοιτάξουμε να καταθέσουμε τροπολογίες και εδώ στην Επιτροπή. Κάποτε που ήμουν πρόεδρος από τη Επιτροπή, θυμάμαι ότι το ζήτημα αυτό μας απασχολούσε συνέχεια στην ημερήσια διάταξη και λέγαμε συνέχεια ότι αν δεν έχουμε τα κείμενα αυτά τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν για να τα κοιτάξουν οι συγητές, πολύ απλά θα τα απορρίπτουμε εκ των προτέρων και αυτόματα. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο αποτελεσματικό από το θέμα τη ονομαστικής κλίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριο Γκάιερ. Ναι, κοιτάξτε. Να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο αξιότιμο κύριο Δεπρέ. Ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου υπάγεται στο τμήμα 5, τμήμα 5 της, ε, του προπολογισμού. Αυτό το τμήμα 5 υπάγεται στους κανόνες για την προπολογισμό. Άρα, το Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει ότι, ε, για παράδειγμα, δεν ε, συμφωνούμε με το χύψη έξοδο του Κοινοβουλίου. Δεν το κάνει όμως αυτό. Υπάρχει μια συμφωνία κυριών. Ότι δεν θα σας πειράξουμε τον προπολογισμό μας, μη μας πειράξετε και εσείς το δικό μας. στα πλαίσια της απαλλαγής δηλαδή. Έχει αυτό μία κάποια λογική. Δεν συμφωνώ, το λέω ξεκάθαρα, δεν συμφωνώ με τη λογική αυτή. Απλά την υπογραμμίζω για να μην βρεθούμε σε κατάσταση όπου θα ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία από το Συμβούλιο θα ερμηνευτεί ως πρόσκληση να αναμειγνύεται στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν θα το θέλα σε καμία περίπτωση. Η διαδικασία του προπολογισμού έχει ως έχει. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ε, διαδικασία αυτή στα πλαίσια του Κοινοβουλίου, αλλά θα ήθελα να σας επισημάνω ότι υπάρχει και δεύτερη αρχή προϋπολογισμού, η οποία ενδεχομένω να το πάρει αυτό ως πρόσκληση να αναμειχθεί. Γιατί αυτό θα έχει την εξή συνέπεια μάλλον θα έχει τις συνέπειες τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε. Ο Ευχαριστώ να επαναλάβω ότι αυτό που συζητάμε δεν είναι και καμία κοσμογονική αλλαγή. Θεωρώ όμως ότι είναι θετική η προσέγγιση μας. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας μας έχει κάνει σύνομο θέτη. Δεν είμαστε κοινοβούλιο με πλήρης αρμοδιότητες κοινοβουλίου βεβαίως. Άρα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Ποιος αποφασίζει γιατί και πότε. Πρέπει να το επιτύχουμε αυτό και οι προτάσεις του Προέδρου πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα Ίσως και αυτοί, και αυτή οι κύριοι της Συμφωνίας Κυρίων ε, του 70 να ήταν υπέρ λίγο περισσότερες σαφήνειας αλλά μάλλον ε, δεν κυκλοφορούν πλέον. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο κ. Γκάιρ. Να προσέξουμε δηλαδή να μην έχουμε προβλήματα συμπεριφοράς των μεν προς τους δε. Αλλά τίθεται το ερώτημα. Υπάρχει κάτι στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου ή γενικότερα για το οποίο ντρεπόμαστε. Αν υπάρχει, ας ανοίξουμε αυτό το κουτί της Πανδώρας. Ας παρεύουμε και στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Γιατί είμαστε το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα διαφάνειας, αλλά είμαστε παρόλα αυτά πολύ διαφανείς. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, δεν είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις των Επιτροπών. Δεν μπορεί να πάει κανείς. Ούτε και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να μάθει πώς ψηφίζει ο καθένας. Και κανείς στη Γερμανία δεν θεωρεί ότι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Κανείς δεν μοιάζει να ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει. Κατά την τελευταία συζήτηση για τον εσωτερικό κανονισμό επιβάλαμε οι τελικές ψηφοφορίες να είναι ονομαστικές. Καλό είναι αυτό. Και θέλω να πω ότι εάν με τέτοια επιδεικτική συμπεριφορά θα απομακρυνθούμε η μεν εκ των δε, τότε αυτό δεν μπορεί να είναι θετικό. Βεβαίως είναι καλή η διαφάνεια, αλλά να μην επιμένουμε συνέχεια. Βεβαίως μπορούμε να βελτιώσουμε ορισμένα θέματα, αυτό είναι σαφές. Αυτό που επέκρινε ο Πρόεδρος είναι ότι μια μάχη που χάσαμε ε, τη χάσαμε γιατί επιμείναμε πολύ σε τροποποίηση των ε, προτάσεων του Προεδρείου. για το Συμβούλιο. Γένς, για πρώτη φορά το Συμβούλιο κινείται και όμως κινείται για να χρησιμοποιήσω αυτή τη διατύπωση του Γαλιλαίου. Μας έστειλε ορισμένες εκθέσεις στο Συμβούλιο των γενικών του διευθυντών. Δηλαδή, στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής του Συμβουλίου έχουμε επιτύχει βελτιώσεις. Βλέπω βέβαια τι περιέχεται και τι δεν περιέχεται στα έγγραφα που μας στέλνουν και τι θα θέλαμε και κατόπιν επανερχόμεθα έναντι του Συμβουλίου και ζητάμε περισσότερα. Και επιτύχαμε εκπληκτικές βελτιώσεις, σημαντικές Η συνθήκη της Λισαβόνας βέβαια αποδυνάμωσε την Επιτροπή μας, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο διαπραγματεύθηκαν ε, οι συνάδελφοί μας. Οπωσδήποτε υπάρχουν διατάξεις που ισχύουν εδώ και 60 χρόνια και που πρέπει να προσαρμοστούν. Εκεί λέγεται ότι το Κοινοβούλιο δίνει απαλλαγή μόνο για τον προπολογισμό της Επιτροπής. Γιατί όταν ιδρύθηκε υπήρχε μόνο ο προπολογισμό της Επιτροπής. Και όλα τα άλλα τμήματα που είναι τώρα εκτός του προπολογισμού της Επιτροπής τότε ήταν εντός. Ε, εν τω μεταξύ εμείς αναπτύξαμε τη δική μας δίκηση αλλά δεν έγιναν οι αναγκαίες αλλαγές. και ορισμένες φορές μας λέει γραμματεία του Συμβουλίου του ούτως ή άλλως ε, δρούμε παράνομα. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φοβόμαστε ότι εκ των υστέρων το Συμβούλιο θα αναμειχθεί στην ε, απαλλαγή του ε, Κοινοβουλίου γιατί δεν το προβλέπουν οι συνθήκες. Ούτε για τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει απαλλαγή. Θα ήθελα να υπήρχε μεγαλύτερη ευαισθησία για το θέμα αυτό αλλά για μένα οι ονομαστικές ψηφοφορίες δεν είναι τόσο σημαντικό. Για παράδειγμα, εάν ορισμένοι καταλάβαιναν τι σημαίνει αυτή η αυστηροποίηση του κανόνα διεντολογίας των επιτρόπων, τότε θα το είχαν ψηφίσει, πιστεύω. Φτάσαμε στο τέλο αυτή τη ανταλλαγή απόψεων που πήγε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πραγματικά εκφράζω την ικανοποίησή μου που σε τόσο λίγο χρόνο ε, βρήκαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε αυτέ τι απόψει. Ε, είναι κάποια θέματα που είναι κάπω ε, δυσάρεστα. Είναι απογοητευτικό να είναι κανεί στην Επιτροπή Πολιτισμού να κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και μετά στην Ολομέλεια να ακούει το Γενικό Γραμματέα να απευθύνει έκκληση αντίθετη με όσα έχουν υπερψηφιστεί εδώ. Κάποιε φορέ καλό είναι να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι θεμελιώδει κανόνε. Πρέπει να γινόμαστε και λίγο σεβαστοί. Να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά που κάνουμε εδώ έχουν και κάποιο νόημα. Και κάποιο λόγο ύπαρξη. Εάν μιλούμε λοιπόν για επενδύσεις και θέλουμε να τις διαχωρίσουμε με κάποιες μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες, αυτό είναι γιατί σήμερα δεν έχουμε καμία πρόπτικη προς στιγμή. Ο προπολογισμό που εγκρίνουμε και για να υπάρχουν αρκετές πιστώσεις ε, που δεν έχουν ε, ε, θα πανηθεί στο τέλο τη χρονιά, τι θα γίνει, θα τα παίρνουμε αυτά για να χρηματοδοτούμε νέα κτίρια, τι νόημα έχει. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το αποδεχτούμε αυτό, με συγχωρείτε συνάδελφοι, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορεί ένα θεσμικό όργανο να δέχεται αυτό το είδο τη λειτουργία. Επιμένω λοιπόν επ' αυτού και η απάντηση που έλαβα χθε από τον Γενικό Γραμματέα είναι πραγματικά νομίζω τελείω ε, άστοχη. Διότι μα λέει δεν ξέρω τι συνέπειε θα υπάρχουν, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ε, ποιο είναι το θεσμικό όργανο που μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά είναι κάτι που μας φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, σε ό,τι αφορά τις ονομαστικές ψηφοφορίες. Όντως, πήγατε τη βαλίτσα λίγο μακριά. Όμως απευθύνω έκκληση προς όλους του συναδέλφους που παίρνουν μέρο στο Προεδρείο. Να είμαστε απαιτητικοί. Ναι, με ενδιαφέρει και από την πλευρά της Γαλλίας. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα παρλαμεντάριο στο Παρίσι, λέει. Γιατί για ποιο λόγο. Πότε το αποφασίσαμε ε, και πότε το συζητήσαμε. Κάποια μέλη του Προεδρείου λέει ενδιαφέρονταν και ωραία, θα το κάνουμε. Τι είναι αυτό, ε, ε, δαπάνη λειτουργία που έχει λόγο για τον υποθεματικό ρόλο που θέλουμε να αναλάβει στην όλη της ε, διαχείριση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Τέλο πάντων, τι γίνεται με το Συμβούλιο ουσιαστικά. Δεν ε, κοιτάζει τι δικέ μου, του δικού μου του λογαριασμού και εγώ δεν μπαίνω στα δικά σου τα χωράφια. Αυτό είναι η ουσία. Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προοδεύσουμε. Τουλάχιστον εγώ δεν αντιλαμβάνομαι έτσι τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Δεν θα πάω μακρύτερα. Ξέρετε ότι οι τροπολογίε πρέπει να υποβληθούν πριν από τι 4 Οκτωβρίου στι 3 το μεσημέρι. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι, ε, τέλο πάντων, αφού έχουμε την ευκαιρία, να συζητήσουμε μεταξύ μα και μετά βλέπουμε τι πορεία θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή, κάποιε αρχέ διοντολογικέ πρέπει να μπορούμε να τι ακολουθήσουμε. Ασχέτω των κανόνων, να ξέρουμε τουλάχιστον ποιο κάνει τι και ποιο έχει ευθύνη. Σα ευχαριστώ για τι αντιδράσει σα. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσε και πολλά υποσχόμενε. Και κύριε Φερνάντε, θέλετε να μα παρουσιάσετε το σχέδιο διορθωτικού υπαριθμών 4 για το 2016. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να σα υποβάλω και να σα παρουσιάσω κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υφίσταται. Δεν μπορώ να σα το παρουσιάσω. Όχι, δεν μπορώ να σα ε, παρουσιάσω το διευθυντικό σχέδιο προπολογισμού παριθμού 4. Δεν, έχει, δεν το έχουμε παραλάβει, δεν ε, ε, υφίσταται ακόμη. Η Επιτροπή νομίζω δεν είναι εδώ. Εάν ήταν, θα τη ρώταγα πότε θα λάβουμε το διευθυντικό υπαριθμό 4 Ποια είναι τα στοιχεία που θα μπορούσαμε να περιμένουμε να υπάρχουν στο σχέδιο αυτό προπολογισμού, το διευθυντικό υπαριθμό 4, αν είναι χρήμα που θα επιστρέψει ε, μέσα από τις καθ, καθυστερήσεις λόγω ε, πλημελούς ε, εφαρμογής, και εκταμείευση, εάν είναι ε, ε, σχετιζόμενο με το, αν αυτό το θέμα σχετίζεται μάλλον με, το, με την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, τι θα γίνει με την επαναπροσαρμογή των στόχων μα, αυτέ τι ερωτήσει θα μπορούσα να τι θέσω για να τροφοδοτήσω τη συζήτηση, αλλά το σχέδιο δεν υπάρχει. Το υπαριθμό 4, το διαδοτικό 4 δεν υπάρχει. Πρόεδρο, κερδίζουμε χρόνο έτσι. Η κυρία Γεωργίευα νομίζω όμω ότι ασχολείται και δεν θα φύγει τόσο εύκολα εάν ε, δεν δώσει μορφή σε αυτό το διευθυντικό Νομίζω πρώτα θα το κάνει το διευθυντικό υπαριθμό 4 να υπάρξει και μετά θα φύγει. Η υπαριθμό 15 έκθεση αναβάλλεται. Ο κύριος Όλμπριχτ τώρα. Για τις διατάξεις που θα μπορούσαν να προβλεφθούν για να παράσχουμε βοήθεια και συνδρομή σε κάποια κράτη. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πρόκειται για την γνωμοδότηση για το πρόγραμμα στήριξη διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. Μια νέα ιδέα που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος το οποίο θα ενισχύσει τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις στα κρατημέλη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα, πρόγραμμα, ένα καινούργιο πρόγραμμα α, τεχνικής αραγωγής για να περάσουν οι διοικητικές, θεσμικές ε, και λοιπές ε, μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Κοιτάμε τις συστάσεις αναχώρα χώρα και θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι πόροι τα κονδύλια θα προέλθουν από την πολιτική συνοχή. Και αυτό αναφέρεται στον προϋπολογισμό. Θα είναι μια νέα γραμμή στην πολιτική συνοχή. Θα είναι τεχνική ρογή όμω. Και θα περάσει από τη Γενική Γραμματεία. Και σκοπός θα είναι, όπως σας είπα, να δοθεί κίνητρο στα κρατημέλη. Και το πραγματικό ζήτημα, η πραγματική πρόκληση είναι ότι το εργαλείο αυτό είναι θελοντικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Προτείνεται απλά στα κράτη-μέλη από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, εκ παραλλήλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη για να ε, πιστήσει την προσοχή στις συστάσεις αναχώρα. Άρα, αποτελεί ένα βήμα για την χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό προβλέπατε για την περίοδο 2017-2020 από πλευράς προϋπολογισμού. 142,8 χιλιάδες. Ε, ευρώ για το 2017 και το μέχρι το 2020 από την πολιτική συνοχή όπως σας είπα και από την 30.000 από την ανάπτυξη της Πέτρου. Τρεις γραμμές προπολογισμού θα χρειαστούν. Δύο στο 1β και μία στο 2, στην, στο τμήμα 2. Και έτσι θα υπάρχει δυνατότητα συμβολή στον οικονομικό αυτό φάκελο από, τον εθνικό, από τους εθνικούς πόρους. Και ξέρουμε ε, ότι γίνονται συζητήσεις από πλευράς των κρατών μελών. Δηλαδή, αν ζητηθεί βοήθεια από το κράτος μέλος και τους χορηγηθεί αυτή η αρρωγή, θα χρησιμοποιηθούν και οι εθνικοί πόροι στο ίδιο παλάθι αυτό στην πρότασή μου υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξουν σε ό,τι αφορά το τελικό κείμενο της έκθεσης. Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το νέο αυτό εργαλείο αποτελεί μόνο ένα τμήμα της ε, λύσης. Δεν πρόκειται από μόνο του να τα επιλύσει όλα, ούτε θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Αν ε, υπάρξει παράταση του προγράμματος ΔΕ μετά το 2020, καλά θα κάνουμε να υπάρξουν νέες γραμμές, όχι να φέρουν τα κονδύλια αυτά από το Ταμείο Συνοχής. Πρόκειται για μια πρόταση ad hoc, όπου χρησιμοποιούμε χρήματα από την πολιτική συνοχής. Και θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να είναι μία μόνο λύση αυτή και οποιαδήποτε παράταση να προαπαιτεί ξεχωριστά κονδύλια στο μέλλον. Δεύτερο στοιχείο. Τα αιτήσια ποσά. Τα ετήσια ποσά θα πρέπει σίγουρα να ελέγχονται και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στην ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού. Θα ήθελα επίσης να ενισχυθεί η αξιολόγηση και ο έλεγχος του συνολικού προγράμματος και να διευκρινιστεί ότι περιλαμβάνονται από σε αυτά στις τρέχουσες τιμές. Αυτό δεν είναι αρκετά σαφές από το κείμενο. Και επίσης η Επιτροπή προτείνει συγχρηματοδότηση, συντελεστή συγχρηματοδότηση 100%. Εγώ θα ήθελα να είναι μέχρι 100%, όχι 100%. Ε, μέχρι 100%. και αναφέρεται ότι πρόκειται για μια τεχνική μετατόπιση μεταξύ των άρθρων σε ό,τι αφορά τις δράσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά τα θέματα οικονομικού φακέλου μέχρι τα θέματα νομιμότητας και υποψηφιότητα. Η νέα πρόταση έχει ως σκοπό να δώσει κίνητο στα κράτη-μέλη να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις, να εφαρμόσουν τις συστάσεις χώρα και τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από την πολιτική συνοχή. Αυτή ήταν λοιπόν η γνωμοδότησή μου και με χαρά να λάβω και τις τροπολογίες σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Όρμπιχτ. Οι τροπολογίες θα πρέπει να επιβληθούν μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 9 ή 10 Νοεμβρίου η Ρέτζη θα ψηφίσει στις 29 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Και τώρα ποιος θα ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλο ο κύριος Μακάου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Συμφωνώ με τις τροπολογίες του. Ο κύριος στόχος των οποίων όπως και του προγράμματος, είναι η βελτίωση του διοικητικού δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις χώρες που ζητούν βοήθεια. Ένα κράτος όταν ζητάει χρήση των πόρων αυτών πρέπει να έχει τις τοπικές και περιφερειακές δυνατότητες για να λάβει τη χρηματοδότηση. Πρέπει να συμμετάσχουν λοιπόν και οι διοικήσεις αυτές και να είναι διαθέσιμες για να εφαρμόσουν μετά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτική φάση. Πρέπει να γίνει μια αποτίμηση εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου και μάλιστα έγκαιρα για να δούμε αν έχει έννοια. Θεωρώ λοιπόν ότι ότι η εκταμίευση θα είναι κάτι μόνο προσωρινό. Η τεχνική βοήθεια η τεχνική βοήθεια που θα δώσει η Κομισιόν θα βασιστεί και στην πείρα από τη βοήθεια που δόθηκε στην Ελλάδα για παράδειγμα και στην Κύπρο γενικά στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αποτίμηση αυτών των προσπαθειών. Πρέπει να εξαγάγουμε τα διδάγματα για παράδειγμα, πώς ε, εκταμιεύθηκαν τα προγράμματα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Επέτυχαν μεν αυτά τα προγράμματα, αλλά δεν ήταν συστηματική η εποπτεία της εφαρμογής των προγραμμάτων. Και γι' αυτό το λόγο να κάνω δύο συστάσεις. Πρώτον, πρέπει να έχουμε σαφή στρατηγική με σαφείς στόχους και προτεραιότητες. Η Κομισιόν πρέπει να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της τεχνικής βοήθειας ελέγχεται, αποτιμάται σε σχέση με τους στόχους ακριβώς του προγράμματος. Αυτή η αποτίμηση πρέπει να είναι συστατικό της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ο Μαραγάλ, ο κύριος Μαραγάλ. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Δεν υπάρχουν αποκλήσει μεταξύ αυτών που είπατε και είναι στο κείμενό σας το αρχικό. Υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες, ίσως να μην είχατε χρόνο μέχρι τώρα να τις εξετάσετε, άρα δεν πρόκειται τώρα να τις παρουσιάσω. Μία γενική όμως παρατήρηση. Το θέμα αυτό δεν είναι καθαρά τεχνικό ή διοικητικό. Δεν είναι δημοσιονομικό μόνο. Είναι ένα σημαντικό τμήμα αυτή η στήριξη στις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που συμπίπτει με πήγουσες ανάγκες και έχει ε, προφανή σχέση με την έννοια των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων. Τι ακριβώς είναι οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, ποια αιρεσιμότητα πρέπει να υπάρχει. Είναι πολύ σημαντική συζήτηση. Ο ρόλος μας πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία αυτών των προγραμμάτων στήριξης. Να μην χρησιμοποιείται αυτό το μέσο όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις επί της ουσίας της υπόθεσης. Αυτή είναι και η έννοια των τροπολογιών μας, ότι πρέπει να είναι από τη βάση προς τα πάνω η κατάρτιση αυτών των προγραμμάτων για να έχουν υποστήριξη. Άρα δεν πρέπει να υποβάλλεται φυσικά απλώς και με θελούσιο χαρακτήρα έτοιμα από το κράτος μέλος. Πρέπει να υπάρχει μια κάποια εγγύηση ότι υπάρχει αποδοχή του αιτήματο αυτού από την κοινωνία, ότι έχει υπάρξει διαβούλευση με τις τοπικές αρχές, με την κοινωνία των πολιτών. Να έχουν δηλαδή προκαθοριστεί ποιες είναι οι ανάγκες, που πρέπει να υπάρξει στήριξη, που θα έχει έννοια να δοθεί στήριξη από την Κομισιόν. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε περισσότερο σε αυτή την προσέγγιση. Και αυτό θα κάνουμε μέσω των τροπολογιών που είναι εδώ στη διάθεσή σας. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω θέλει κανεί άλλο το λόγο. Α, η κυρία Γκρέσλε. Ε, κύριε Σιγητά, να μιλήσει πρώτα ο η κυρία Γκρέσλε. Μου προκαλεί εντύπωση το μικρό, ο μικρός φάκελος. Ε, τι θα καταφέρουμε να καλύψουμε, ο κύριος Αλμπρίχτη. Με προκάλεσε η κυρία Γκρέσλε να αφήσω το δημοσιονομικό σκέλος και να μιλήσω πολιτικός. Ε, πολιτικός πώ, Το θέμα λοιπόν για μα είναι το εξή. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν διεξαγάγουν τι ε, μεταρρυθμίσει μεταρρυθμίσεις, για ποιο λόγο. Επειδή δεν έχουν χρήματα ή μήπω δεν θέλουν απλά να τις προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις ή μήπω δεν είναι έτοιμα να τις εκτελέσουν. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Εξ όσων καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκοπός είναι να δοθεί κίνητρο στα κράτη-μέλη να κάνουν τι μεταρρυθμίσεις αυτές. Φυσικά τα χρήματα δεν είναι πάρα πολλά και δεν ε, ε, θα επιτρέψουν να γίνουν πραγματικά, πραγματικές μεταρρυθμίσει. μεταρρυθμίσεις. Αλλά το, πραγματικά, το πραγματικό πολιτικό ερώτημα το οποίο έχω θέσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώς σκοπεύετε να δώσετε κίνητο στα κράτη-μέλη να ζητήσουν χρήματα. Γιατί είναι σε βάση. Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλουμε να εκτελεστούν οι συστάσει σε ένα χώρα, δεν υπάρχει περιθώριο. Θα πρέπει να ζητηθούν τα κονδύλια αυτά για να εφαρμοστούν οι διαθροτικέ μεταρρυθμίσει. Είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι τα πραγματικά χρήματα αυτά για την εκτέλεση των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν νομίζω ότι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος τα 140.000 ευρώ έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Είναι συμβολικό ποσό. Εξαρτάται φυσικά και από την περίπτωση. Αυτό λοιπόν προέρχεται ως παράδειγμα από την Ελλάδα. Μάθαμε από την Ελλάδα και σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο οικονομικό. Συμφωνώ όμως ότι είναι μικρό το ποσό. Αυτό είναι ο πολιτικός ε, λοιπόν τρόπος σκέψης. Ας το προσπαθήσουμε. Αλλά α μην λέμε ότι δίνουμε χρήματα για διδακτικέ μεταρρυθμίσει, γιατί δεν στέκει κάτι τέτοιο. Bien. Nous voici arrivés au terme de nos travaux. Ωραία. Ε, φτάσαμε στο τέλος των εργασιών μας. Ευχαριστώ τους εισηγητές. Ευχαριστώ όσους μείνατε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ε, διάφορα. Έχει κάνει τίποτα στα διάφορα. Όχι. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει συνεδρίαση για αύριο το πρωί, αλλά ε, εξαντλήσαμε την σε διάταξη, οπότε δεν θα συνεδριάσουμε αύριο το πρωί και οι επόμενη συνεδριάσεις θα είναι 10 ε, και 11 Οκτωβρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Λήξη της συνεδρίας.